Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Καταρχήν μια ανακοίνωση. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τα κείμενα τα οποία με σε ε, υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο θα θεωρείται ότι εγκρίνονται αν μέχρι 24 ώρες προθεσμίας από μια κοινοβουλευτική ομάδα ή από ευρωβουλευτές δεν δηλωθεί ότι ζητείται να τεθούν υποψήφιση. Είναι και στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης θα εμφαίνονται. Σαν επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κοινή συζήτηση για το θέμα της δικαιοσύνης και αφενός για την έκθεση Berlinguer πρόγραμμα δικαιοσύνη 2014-2020 και την έκθεση Göns, πρόγραμμα δικαιώματα και ηθαγένεια 2014-2020 θα ξεκινήσουν οι συγητές και ξεκινά ο κύριος Berlinguer, έχει τέσσερα λεπτά παρακαλώ Grazie, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός τον οποίο καλούμεθα να εγκρίνουμε σήμερα αφορά στο επταετές πρόγραμμα παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης.